Παρακαλώ πάρτε θέσεις για να έχω τουλάχιστον την εντύπωση ότι έχουμε αρχίσει τις εργασίες μας. Λοιπόν, στη γνωμοδότηση που σας προτείνω αναφέρω ότι η Δημοσιονομική Επιτροπή καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων που είναι υπεύθυνε, που είναι αρμόδιε επί της να ενσωματώσουν το σχέδιο ψηφίσματός μας στην δική τους πρόταση ψηφίσματος. Θέλουμε να προσθέσουμε τα εξής. Καταρχήν μια διαπίστωση. Οι συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πολιτικές εξελίξεις μας οδηγούν στο να σκεφτούμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Είτε αυτές αφορούν το ΝΑΤΟ, είτε αυτές αφορούν ε, την αμερικανική βούληση παρέμβασης ε, σε σχέση με το παρελθόν. Επήγει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση Άμυνας. Βεβαίως οι οικονομικοί πόροι εδώ παίζουν ένα ρόλο κλειδί και αν πάμε προς μηχανισμούς ε, όπου θα μοιραζόμαστε ε, τα έξοδα, θα μοιραζόμαστε ε, τις δαπάνες και το κόστος, αυτό θα ήταν εξαιρετικά θετικό, διότι το κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα της ασφάλισης και της άμυνας μας κοστίζει 26 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, διότι έχουμε επικαλύψεις, διότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ε, σε ό,τι αφορά ε, τις δημόσιες προμήθειες η χρησιμοποίηση κοντιλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα του προπολογισμού της θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα συνοχής και αλληλεγγύης και θα μας επέτρεπε μια πιο διαφανή, ένα πιο διαφανή έλεγχο της χρηματοδότησης. Χρειάζεται τα εξή στάδια. Πρώτα, διεύρυνση και μεταρρύθμιση του μηχανισμού Αθηνά για την κατανομή των βαρών, για να έχουμε μια πιο συλλογική χρηματοδότηση των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θέσπιση μιας μόνιμης διαρθρωτικής συνεργασίας, ΠΕΣΚΟ, όπως βλέπετε στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξεπάγωμα του κονδυλίου για τον προπολογισμό της ε, Ένωσης Άμυνας, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, και οι, πρω... οι πρώτες δράσεις ε, είναι ένα καλό βήμα. Πριν από ε, μια εβδομάδα ψηφίσαμε το πρώτο, την πρώτη δόση των 25 εκατομμυρίων. Ελπίζουμε γρήγορα τα κράτη-μέλη να βρουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Τώρα, πιο μακροπρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να σκεφτεί πώς θα έχει ένα κοινό προπολογισμό για να χρηματοδοτήσει τον πυρήνα των ε, ενσωματωμένων στρατιωτικών δυνάμεων της Ένωσης, να υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό έρευνας ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από νέα κονδύλια, από επιπλέον κονδύλια δηλαδή χαιρετίζω την παρουσία του κυρίου Ντόνζο στον οποίο την ευθύσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ε, για την ε, ε, τις κεντρικές γραμμές της γνώμης σας. Βεβαίως υπάρχει δυστυχώ αυτή η πίεση από τα διεθνή γεγονότα, από τι διεθνείς εξελίξεις και αρχίζουμε και εμεί ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να σκεφτόμαστε πιο σοβαρά τι ευθύνε που μα αναλογούν ω Ευρωπαίοι για να εξασφαλίσουμε τη δική μα ασφάλεια, να μην εξαρτώμαστε πάντα από άλλου. Γι' αυτό λοιπόν στην γνωμοδότηση που συντάξατε θα ήθελα να επανέλθει ο όρος στρατηγική αυτονομία ε, που αποτελεί πλέον μέρος ε, της φρασιολογίας στα κείμενα του Συμβουλίου. Ε, εδώ και καιρό υπήρχε στα κείμενα του Κοινοβουλίου, τώρα ε, υπάρχει και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Σε σχέση με αυτά που επενθυμίσατε, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιμείνουμε στο γεγονός ότι έχουμε στη διάθεσή μας τα εργαλεία που χρειαζόμαστε στα πλαίσια τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έχει βεβαίω εμπλουτιστεί η συνθήκη τη Λισαβόνα από κάποιε δημοσιονομικέ ε, δράσει, ε, όπω οι προπαρασκευαστικέ ε, δράσει, ε, αλλά τα εργαλεία, τα μέσα, τα θεσμικά και τα νομικά υπάρχουν στη συνθήκη τη Λισαβόνα, απλώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Εδώ και χρόνια εγκρίνουμε κείμενα ε, στις επιτροπές μας ζητούμε την ρητή, την αυστηρή εφαρμογή της θήκης Λισαβόνας. Έχω δύο μικρές επιφυλάξεις σχέση με το κείμενο που μας προτείνατε. Είμαι κάπως επιφυλακτικός ε, σε ό,τι αφορά το κόστος της μη Ευρώπης. Διάβασα προσεκτικά την έκθεση που αποτελεί τη βάση αυτής της ε, αξιολόγησης και δεν έχω πιστεί για ε, την δημοσιονομική εγκυρότητα αυτού του κόστου της μη Ευρώπης, γιατί είναι στο μέσο που δεν υπήρξε ποτέ Ευρώπη. Αυτές οι προβολές λοιπόν που κάνετε δεν λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από ιδιαιτερότητες στον τομέα της άμυνας. Παραδείγματο χάρη, το βασικό κόστο τη μη Ευρώπη είναι όταν τα δύο τρίτα των χωρών τη Ένωση, που όταν πρέπει να επιλέξουν εξοπλισμό ευρωπαϊκό ή αμερικανικό, αγοράζουν αμερικανικό εξοπλισμό. Αυτό είναι κόστο μη Ευρώπη. Αλλά δεν ποσοτικοποιείται αυτό στην έκθεση. Ενώ η απόφαση ενό κράτου μέλου πρόσφατα ε, μπορεί να διακυβεύσει το μέλλον της Ερμπάς. Ε, δηλαδή το, η έννοια του κόστου της μη Ευρώπης είναι δύσκολο ε, να ποσοτικοποιηθεί ε, και να εντοπιστεί. Οπότε δεν θα, δεν θα επέμενα στο επιχείρημα αυτό. Να πούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν μια σειρά από κοινές ε, ε, ενός μοιράσματος των ε, πόρων στην αρχή της διαδικασίας. Τώρα, γίνεται αναφορά στην ολοκληρωμένη ε, στρατιωτική δύναμη. Ε, όταν μιλάμε για επιχειρησιακές μονάδες, για μονάδες μάχημες δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορούμε στην Ευρώπη με βάση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων να έχουμε ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη στρατιωτική δύναμη. Διότι εκεί χρειάζονται κανόνες ε, για, την, ε, για το πώς ε, μπαίνει κάποιος σε ένοπλη κατάσταση, στο, στους όρους εμπλοκής, άλλους όρους εμπλοκής έχει η Γαλλία, άλλους η Γερμανία, κάθε μία έχει παραδόσεις της. Είναι κάπως λοιπόν φιλόδοξο να μιλάμε ήδη από τώρα για ολοκληρωμένη στρατιωτική δύναμη. Αυτά έχω να πω. Είναι μια πολύ καλή βάση το κείμενό σας και συγκλίνω σε πολλά σημεία με αυτά που είπατε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντονζό. Ο κύριος Γκεγέρ έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. να συζητήσω και να σας πω εξ αρχής ότι είμαι λίγο ανήσυχο για αυτά που συζητάμε εδώ. Γιατί στον προπολογισμό για τον οποίο ευθύνομαι εγώ, κάναμε και αποφασίσαμε να υπάρχουν προπαρασκευαστικά μέτρα με κάποια συγκεκριμένα ποσά. Αλλά ήδη από αυτή τη φάση ανέκυψε το ερώτημα το κατά πόσο στον προπολογισμό στις κατηγορίες στις οποίες θέλουμε να λάβει η χώρα αυτή η πλωτική ενέργεια, έχουμε επαρκή ε, κονδύλια για να χρηματοδοτήσουμε. Τα βρήκαμε τα κονδύλια. Και παρατηρώ και με ανησυχεί κάπως αυτό ότι σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποεπιτροπή α, ε, α, ε, για τα θέματα ασφάλειας πάντα βλέπουμε προτάσεις για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και το σκέλος που συνδέεται με τη χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής ε, είναι μάλλον αυθαίρετο, για να το πω και ευγενικά. Το συζητήσαμε επί μακρόν για το πώς η πρόταση του Συμβουλίου για την προετοιμασία του μεσοπρόθεσμου του δημοσιονομικού πλαισίου την αξιολογούμε και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι επιπρόσθετα κονδύλια για μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν διατίθενται στο τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και βλέπουμε από συναδέλφους ε, του Κοινοβουλίου που δεν ασχολούνται καθημερινά με τα θέματα χρηματοδότησης ότι οι αξιώσεις που θέτουν έναντι του προϋπολογισμού είναι εκτενείς. Κύριε Ντανζό, είπατε ότι έχουμε τη δυνατότητα, Ίσως το είπε και ο κ. Αρτουή, θυμάμαι, ο πρόεδρο, ότι ίσως από το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν είναι σαφές όμως πότε, ότι θέλουμε 500 εκατομμύρια για προγράμματα έρευνας. Πολύ απλά σε αυτή τη φάση δεν τα έχουμε τα χρήματα αυτά. Ο κανονισμός για τον ορίζοντα 2020, όπως ε, προτείνεται στην παρούσα φάση, ε, αποκλείει θέματα έρευνα για εξοπλισμό που ζητάτε. Άρα, ή θα πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο ή να περιμένουμε το επόμενο. Και πάλι λοιπόν να το πολιτικό ερώτημα, πολιτικό ερώτημα, πολιτικό ζήτημα. Από τα χρήματα που έχουμε στην πολιτική έρευνα, στα οποία δεν είναι και πάρα πολλά, είμαστε σε θέση να διαθέσουμε 500 εκατομμύρια 10 έως 15% δηλαδή για την έρευνα για τον εξοπλισμό. Όταν η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο αποφασίζουμε ξανά και ξανά ότι αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε είναι η καινοτομία. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί ο εξοπλισμός να είναι καινοτομικό σε κάποια φάση, αλλά στην τελική ανάλυση ένα τεθρακισμένο είναι τεθρακισμένο. Δεν αποτελεί α, επένδυση που θα έχει προστιθέμενη αξία και είμαι πάρα πολύ διστακτικό για το κατά πόσον μπορούμε να παρέμβουμε στον προπολογισμό. Επιπλέον κονδύλια μάλιστα. Εντάξει, να το πούμε ξεκάθαρα. Διατύπωσα και μια τροπολογία για την γνωμοδότησή σα, Πρόεδρε, που τα διευκρινίζει αυτά, γιατί πιστεύω ότι η διατύπωση ότι μόνο στο Ταμείο άμυνας. Χρειαζόμαστε επιπλέον κονδύλια. Επειδή χρειαζόμαστε τα 500 εκατομμύρια, ε, πιστεύω ότι αν συμφωνήσει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου να γίνει ένα κατανομή των 500 εκατομμυρίων αυτών, ε, εντάξει, αλλά εγώ πολιτικά δεν συμφωνώ. Αν το συμφωνήσει το Κοινοβούλιο, εντάξει. Αλλά θα πρέπει και στο Κοινοβούλιο εδώ να προσανατολιστούμε προς την ε, εξής κατεύθυνση. Να μην προβαίνει ο καθένας στην κάθε επιτροπή σε προτάσεις ε, που να ακολουθούν μία λογική του «Α, ζητάμε πάντα παραπάνω από ό,τι ως τώρα, γιατί θέλουμε μία πιο αναπτυγμένη πολιτική άμυνας», αλλά θα ήθελα να ορίσουμε μία σειρά του τι πρέπει να γίνει, ποιε είναι οι προτεραιότητε και ποιο θα πληρώνει όλα αυτά. Γιατί αυτό που ανησυχεί είναι ότι αν το Κοινοβούλιο δεν αποφασίσει εγκαίρω επί συγκεκριμένων θέσεων, θα τα αποφασίσει όλο το Συμβούλιο, όπω συνηθίζει. Και οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, ενδεχομένω να πάρουν τι δικέ του αποφάσει και τι δικέ του προτεραιότητε για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και να μην εισακούσουν απαραίτητα τι επιθυμίε του Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα και στην Επιτροπή μας να καταρτήσω μια έκθεση πρωτοβουλίας για την χρηματοδότηση της μελλοντικής πολιτικής άμυνας. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό αξίζει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω, να καταναλώσουμε λίγο παραπάνω θέα ουσία. Ευχαριστώ. Επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Comment, uh, whereas... Έχω ένα μικρό σχόλιο να κάνω. δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό το οποίο συζητάμε. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη για την ασφάλειά μας. Από την άλλη έχω να κάνω μια πολιτική παρατήρηση. Αν κάποιος από μας ανησυχεί για την σύνδεσή μας με την βορειοατλαντική διάσταση. Εγώ είμαι υπέρ φυσικά αυτού του συνδέσμου. Εφόσον ανησυχούμε γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την ρητορική η οποία θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια. Η κατάσταση έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα στις Ηνωμένε Πολιτείες λίγο εύθραυστη. Δεν θα επιθυμούσαμε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους Αμερικανούς ότι είμαστε διατεθειμένοι εμείς και έτοιμοι να αναλάβουμε τα της ειδική μας ασφάλειας, διότι πολύ απλά δεν είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντονανό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουμε αρκετοί εδώ που πριν από τις ακλογές που έδωσαν τον κύριο Τραμπ είχαμε προειδοποιήσει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες σε σχέση με την ευρωπαϊκή άμυνα. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια κάποια επιθυμία να προχωρήσουμε. Είναι μια καλή πρόταση. Από την άλλη και ο Χανσκέρτ έχει δίκιο, οι πιέσεις οι δημοσιονομικές ε, είναι τεράστιες στα πλαίσια του σημερινού προϋπολογισμού δεν μπορούμε να φανταστούμε την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Ή θα πρέπει να υπάρξουν ήδη οι πόροι ή θα πρέπει να υπάρξουν αμοιβεοποιημένες αν θέλετε οικονομικές συνεισφορές από πλευράς πολλών κρατών. Λοιπόν, να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Μίανμαρ να χαιρετήσω τον πρόεδρό της που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Καλώς ήλθατε συνάδελφοι. Και οι νομικές υποθέσεις και οι δημοσιονομικές υποθέσεις συνδυάζονται προς όφελος των λαών μας. Ε, Λοιπόν, στα πλαίσια τα δημοσιονομικά 14-20 τα προβλήματα αυτά δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται. Αλλά πάντως η συνθήκη της Λιφασμόνας μας δίδει κάποιες δυνατότητες που δεν έχουμε εφαρμόσει μέχρι τώρα. Ο κ. Ντανζουάν, να υπενθυμίσω αν μου επιτρέπετε ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Γκάιερ για τις δημοσιονομικές ανασφάλειες ή αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν το μέλλον. Είναι μια πολύ θεμητή ανησυχία και θα ήταν σωστό να το συζητήσουμε το θέμα αυτό <clears throat> με τον πιο εξαντλητικό τρόπο και να εξετάσουμε και το θέμα των συνεισφορών των κρατών μελών. Θα ήθελα επίσης εδώ να υπογραμμίσω τον κίνδυνο που παρουσιάζει μια ορολογία ολίγων θα έλεγα προκατηλημένη. Μιλάμε δαπάνες στον τομέα της έρευνας. Ε, δεν μιλάμε για αυστηρά στρατιωτικές δαπάνες και δεν μιλάμε για δαπάνες αυστηρά σε σχέση με εξοπλισμούς στρατιωτικούς. Μιλάμε για συστήματα πλοήγησης, σαν παράδειγμα ε, για μη επανδρομένα πτυτικά μέσα Μιλάμε επίσης για ιατρικά συστήματα που θα ήταν χρήσιμα σε χειρουργία εκστρατεία. Είναι μια ολόκληρη σειρά από ερευνητικές δυνατότητες οι οποίες δεν προορίζονται αποκλειστικά στο να γεμίζουν τις τσέπες των εμπόρων που χτίζουν κανόνια. Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με την χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω και εγώ στον κύριο Ντονζόν, να του πω ότι καλό θα είναι να διευκρινίσουμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για στρατηγική αυτονομία ή για αυτονομία στο επίπεδο της στρατηγικής στο σημερινό διεθνές πλαίσιο. Τώρα, για τις επιφυλάξεις τις οποίες εκφράζει στα δύο συγκεκριμένα σημεία θα βρούμε μια διατύπωση για να τις ξεπεράσουμε σχετικά με τον Γιάνς Γκάιγερ. Είναι σαφές ότι στον σημερινό προϋπολογισμό δεν έχουμε τα μέσα τα οποία να είναι στο ύψος των απαιτήσεων που έχουμε. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να προετοιμάσουμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό. Το Συμβούλιο θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό και να προσπαθήσει να προκαταλάβει τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο και για την έρευνα σκέφτομαι ότι και σε άλλες χώρες στα πλαίσια των στρατιωτικών λεγόμενων ερευνητικών προσπαθειών γίνονται βήματα προόδου τα οποία βοηθούν και τους Νομίζω ότι αν βοηθήσουμε την έρευνα στον στρατιωτικό τομέα βοηθάμε την έρευνα γενικότερα και στον μη στρατιωτικό τομέα. Και καλό θα είναι να μην φανούμε διστακτικοί εγώ φυσικά εδώ υπογραμμίζω και συμφωνώ με τις επιφυλάξεις του κυρίου Σαβάρμα και να πω επίσης τον κύριο Ντονανό ότι σε επίπεδο δημοσιονομικό θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε όπως προχωρήσαμε στα πλαίσια της αποκέντρωσης στη Γαλλία. Όταν περάσαμε σαν παράδειγμα στη μεταφορά των πόρων που έδινε στην περιοχή της Λιμόζ η λιμόζη είναι αυτή η οποία τώρα μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα ποσά αυτά εξ αρχής με αυτονομία. Λοιπόν, οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν πριν από τις 16 Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου στην Επιτροπή και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια την 13η Μαρτίου. Λοιπόν, θα σας εγκαταλείψω τώρα. Α, ο κύριος Μάνγκα για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο λέξεις επιτρέψτε μου σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών ε, αμυντικών ε, δραστηριοτήτων. Ενδεχομένως να μην χρειαστούν καν επιπρόσθετοι πόροι. Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων των μονομένων χωρών και ενδεχομένως να κλειτώσουμε έτσι, να εξοικονομήσουμε 35 έως 105 δις ανά έτος. Τεράστιο ποσό. Ναι, υπάρχουν ε, ενιαία κτίρια, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, ε, τρίτες χώρες, ε, όπου βρίσκονται μαζί αντιπροσωπείες των χωρών της Ένωσης. Έτσι μπορούμε να εξοικονομήσουμε ε, στο ίδιο κτίριο να συνεπάρχουν ε, διάφορες χώρες και έτσι ε, δεν θα μας κατηγορούν για διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Αλλάζει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να προχωρήσουμε. Το επόμενο σημείο στην μέσα διάταξη έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για, την, για το πολιτικό συντονισμό της Ένωσης, την ετήσια έκθεση του 2017. Ο κ. Ντενανό είναι, είναι ο εισηγητής. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αυτό. Αυτή η έκθεση βεβαίως ε, ε, είναι κάπως ε, εσπεσμένη, αλλά υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Το θέμα της οικονομικής ανάκαμψης είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πιέσει έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τα μέσα στη διάθεσή της έτσι ώστε αυτή η οικονομική ανάπτυξη να μπορέσει να προχωρήσει. Στην έκθεση αυτή ήθελα να υπενθυμίσω τη σημασία ενός ε, ε, ισχυρού προπολογισμού, ιδιαίτερα μετά τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ανακουφίσουμε και τους εθνικούς προπολογισμού και να χρησιμοποιήσουμε κοινού πόρους. Σε ό,τι αφορά τον, τους μηχανισμούς σταθερότητας, κανείς βεβαίως δεν μπορεί να αντιταχθεί στον μηχανισμό σταθερότητας. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί, αλλά κάποια πράγματα όπως το, το, το, το διεθνή συνεργασία, εδαφική ε, ισορροπία, η συνύπαρξη, θα μπορούσαμε εκεί τα, τα κριτήρια σύγκλησης κάπως να τα ε, σχετικοποιήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα τελωνιακά ε, στους δεσμούς, εδώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ε, για να αποφύγουμε την απάτη της ΦΠΑ Πρέπει να δημιουργήσουμε όλες τους απαραίτητου μηχανισμούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φορολογική απάτη γενικότερα. Μάθαμε πρόσφατα ότι 172 ε, νέοι ε, ε φορείς ε, φορολογικής ε, παρανομίας ε, έχουν δει στο Λουξεμβούργο μετά τα LuxLeaks και αυτό πραγματικά πρέπει να μας ανησυχεί. Στον τομέα της ανάπτυξης η ανάπτυξη είναι ισχνή για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Και ο βασικό μα στόχο είναι να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση για να δώσουμε προοπτική στου νέου μα. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε περισσότερο τι δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει και τα δύο και να δώσουμε τη δυνατότητα στι μικρέ επιχειρήσει να παίξουν το ρόλο του στον οικονομικό κόσμο. Επίσης θεωρώ ότι ο έλεγχος ο νομισματικός ε, είναι σημαντικός ε, για την οικονομική ανάπτυξη. Ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Επίσης ε, κάτι άλλο που μας κινητοποίησε ιδιαίτερα είναι το θέμα των διαθροτικών ταμείων και οι μακροοικονομικές συνθήκες για την κατανομή των δημοσιονομικών ταμείων, των διαθροτικών ταμείων, συγγνώμη, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε μακροοικονομικά κριτήρια ίσχυσε για την Ισπανία, για την Πορτογαλία. Ε, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, ε, πρέπει να ισχύσει και για άλλους αυτή η ευελιξία. Υπάρχουν λύσεις σε επίπεδο ευρωζώνης τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε. Είμαι διατηθειμένος βεβαίω να ακούσω τις τροπολογίες που θα υποβληθούν και νομίζω ότι η Επιτροπή μας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε τον κύριο Τενανό και το να ακούσουμε τους συναντέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο για ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αιτήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη για το 2017 τονίζει τις βασικές οικονομικές προτεραιότητες της Ένωσης και δίνει οδηγίε και κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για τα επόμενα χρόνια βάσει τη στρατηγική ε, σε τρεις βασικούς τομείς. Ε, επενδύσεις, συνταγματικέ μεταρρυθμίσεις και χρηματοοικονομική πειθαρχία. Και αναφέρονται λοιπόν εδώ πέρα κάποια θετικά σημεία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει των οποίων μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα στο δεύτερο ημίση του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται σωστά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη αυτή, είναι μάλλον περιορισμένη και μετριοπαθή, σε πιο χαμηλή από ό,τι αναμενόταν και αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω λόγω διάφορων ε, φορέων, δημογραφικές αλλαγές, η τιμή της ενέργειας που αυξάνεται και διάφορες τέτοιες αρνητικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. και της ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεν καλύπτονται όλα τα μακροοικονομικά σκέλη και μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε κάποια ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση του σχεδίου είναι θετική και τα αποτελέσματα είναι θετικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιάρθρωση γιατί στην παρούσα φάση και υπό το μορφότυπο αυτό δεν μπορεί να εγγυηθεί τη μακροοικονομική οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και να ωφεληθούν όλα τα κρατημέλη στη τελική ανάλυση. Κατά δεύτερον, τα αποτελέσματα της μη Συμβατική οικονομική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά τι προσπάθειες που έγιναν, τελικά οδηγούν σε μια περιορισμένη ανάπτυξη των ε, τιμών και ο πληθωρισμός είναι σε προβληματικά επίπεδα. Και το γεγονό ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στα επίπεδα που κινείται λόγω τη προβληματική ε, χρηματοοικονομική πολιτική, θα έπρεπε να μα οδηγήσει ενδεχομένω σε μια αναθεώρηση αυτής κατά τα τέταρτον σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των ε, κεφαλαίων αγορών. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην είναι πλέον καταγερματισμένη η κεφαλαία αγορά στην Ευρώπη και θα πρέπει να είναι πιο ενοποιημένε οι κεφαλαίοι αγορές. Αυτό θα προσελκύσει και θα κινητοποιήσει το κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, για να αντιμετωπίσουμε την ενεργεία των νέων, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ε, εκπαίδευση και στην κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση των νέων στην Ένωση. Προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να έχουν κάποια βασικά προσόντα οι νέοι να έχουν και μια τεχνική διάσταση, όμως και μια επιχειρηματική ικανότητα. Και τέλος, για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, για να αυξηθεί η απασχόληση, θα πρέπει να φροντίσουμε να εξαλείψουμε τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις. Να είναι απλοποιημένο σύγχρονο το φορολογικό σύστημα, να μην αφήνει περιθώρια για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή για να έχουμε επαρκείς πόρους και για τα κρατημέλη αλλά και για την κοινότητα, για την Ένωση στο σύνολό της. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Μάλετιτς. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή και να υπογραμμίσω ότι η ετήσια έκθεση Ανάπτυξη για το 2017 είναι ένα σημαντικό πολιτικό έγγραφο. Αποτελεί και τη βάση ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι ένα σημαντικό έγγραφο το οποίο όλοι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και για τα, στα πλαίσια των εθνικών ε, σχεδίων μεταρρυθμίσεων, τις, συστάσεις αναχώρα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερα από την ετήσια επισκόπηση. Εάν θέλουμε η καινοτόμος Ευρώπη να είναι στην εξηγετικό ρόλο παγκοσμίω, ε, δεν πρέπει να μιλάμε για τα θεωρητικά ταμεία και για δημοσιονομική εξυγίανση και για ενίσχυση επενδύσεων. Εάν δηλαδή συνεχώς έχουμε τις, ε, αναφερόμαστε σε αυτές τις συστάσεις χώρα, αλλά δεν τις εφαρμόζουμε, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι σημαντικό λοιπόν να αλλάξουμε το πώς προσεγγίζουμε ε, και πώς ορίζουμε τελικά αυτήν την ε, ετήσια επισκόπηση. Θα πρέπει να εντοπίσουμε διαρθρωτικά συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες, οι νέοι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς ε, στις χώρες μας. Πολλά τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τις δικές μας ε, ανεπάρκειες και τη δική μας αναπαρτισματικότητα. Παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη ε, στον κόσμο σε ό,τι αφορά την ε, κυκλική οικονομία. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τροποποιήσει τον κανονισμό έτσι ώστε να επιτρέψουμε την διατομιακή συνεργασία και τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Και λόγω αυτού έχουμε αυτή την αργή αντίδραση και άλλοι θα μας προσπεράσουν και οι καινοτόμε ε, επιχειρήσεις μας, όχι μόνο στην κυκλική οικονομία, θα φύγουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε. Σε επίπεδο κρατών μελών ε, είναι πολύ ε, διαφορετικές νομοθεσίες, είναι αυστηροί οι κανόνες, όλα αυτά αποτελούν εμπόδια για την πρόοδο, την καινοτομία, για καινοτόμες λύσεις και βεβαίως και για υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, για να επιλύσουμε λοιπόν αυτές τις δυσκολίες, ε, αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφέστερα σε έγγραφα όπως η αιτήσια επισκόπηση. Και αυτό είναι σημαντικό. Να προσθέσω κάτι για τον κοινωνικό προπολογισμό και το πώς συνδέεται με τους εθνικούς προπολογισμούς. Όταν συζητάμε για το χρέος, όταν μιλάμε μάλλον για αυτό, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει συνέργεια όχι μόνο μεταξύ πολιτικών και διαφόρων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και συνέργειες μεταξύ των προπολογισμών των κρατών μελών, ε, έτσι ώστε ο κοινωνικός προπολογισμό να επιφέρει πραγματικά προσθέμενη αξία, να επιφέρει αλλαγές ε, στα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά σε επίπεδο κρατών μελών, εάν θέλουμε μια πραγματική ενιαία αγορά και καλύτερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις μας, θα πρέπει να κινηθούμε από κοινού και σε επίπεδο προπολογισμών. Το θέμα είναι κατά πόσο εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια τη της επισκόπησης. Ζητούμε κοινέ λύσεις από τα κράτη-μέλη που να είναι ορατές στους εθνικούς προπολογισμού και να συνδέονται, αλλά και, αλλά και να συνδέονται με τον κοινωνικό προπολογισμό. Υπάρχει κάποιο μήνυμα στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2017 για τους εθνικούς προπολογισμού των κρατών Είναι σαφές ε, αυτό για τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια ξαφή επικοινωνία με τα κράτη-μέλη επ' αυτού. Αυτά πρέπει να αναρωτηθούμε και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Εάν όχι, να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι η 9η Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 15 Ιανουαρίου. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές πάλι στα πλαίσια της αιτήσης επισκόπησης της ανάπτυξης. Η συγκήτρια είναι η κυρία Νιριάντα. Ζήτησε να αναβληθεί το θέμα αυτό, οπότε θα προχωρήσουμε θα το εξετάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Και τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Υπάρχει ένα έτοιμα της κυρίας Χόλμαϊρ να εξεταστεί πρώτα η δική της, ε, το δικό της κείμενο. Ξεκινούμε λοιπόν από το σημείο 13. Θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου για την καταχώρηση δεδομένων εισόδου και εξόδου καθώς και άρνηση εισόδου υπηκών τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των όρων πρόσβασης σε αυτό το σύστημα για σκοπούς επιβολής του νόμου. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. So, and this is my first time, so bear with me. I might Πρώτη φορά λοιπόν θα προτρέψω σε ψηφοφορία. Σας παρακαλώ υπομονή δείξτε. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος παρακαλώ. Ενάρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η υπερφημόν 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 32 υπέρ. Κατά. αποχές. Κατά εγκρίνεται. Οι δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 33. Με προφορική τροπολογία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θέλει κάποιος να το διαβάσει? Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Η 5. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Και περνάμε τώρα στις τελογικές σκέψεις. Τροπολογία υπαριθμών 8. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφοφορία unblock. Η 13, 14, 15, 16, 17 και 18. 13 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21. Αποσύρεται. Η τροπολογία 6 και 7. Η 6 και 7 από, από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Δεκαεννέα ψηφι υπέρ, 11 κατά, καμία αποχή, άρα η γνωμοδότηση εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία είναι στο σημείο υπαρθών 9, η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Κομμουνιδά Βαλενσιάνα, αυτοκινητοβιομηχανία στην Ισπανία. Ο κύριος Έστεμπαν Κοζάλης Πόντς είναι ο εισηγητής. Και να ψηφίσουμε τροπολογία υπερθμών 1. Α, συγγνώμη να ξεκινήσουμε με τα άρθρα και να αφήσουμε στο τέλος τα υπόλοιπα. Στην παράγραφο 1, τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές, παρακαλώ, για σηκώνστε καλύτερα τα χέρια σας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Διευκρινίζω ότι κάνουμε μία μικρή αλλαγή στην ε, κατάλογο ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τα άρθρα. Να περάσουμε πρώτα λοιπόν στην ψηφοφορία των άρθρων. Τροπολογία 7, υπέρ. Συγγνώμη.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 και στη συνέχεια να πάμε στα citation στην τροπολογία. So I learned that you have to take this out of the folder. Amendment 11 and, and 12, block vote. Amendment 11 and 12. 11 12 από κοινού. Αυτό νομίζω ότι είναι σαφές. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 13. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 17. Οι 17 και 18 έχουν καλυφθεί. Οι 17 και 19, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Οι 17 και 19 σε κάποιους καταλόγους ψηφοφορίας περιλαμβάνεται, σε κάποιους όλους όχι συμβιβαστική καλύπτει τις 17 και 19. Πιστεύει πιο τη ευρύτερη χρήση της εξαίρεσης για τα όρια για, την, για τους ε, ε, υπαλλήλου τη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δυνατότητε που σχετίζονται με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα πρέπει να εκτιμώνται προσεκτικά και κατά περίπτωση προσπαθώντας να περιοριστεί η στρεβλωμένη χρήση του προϋπολογισμού και θα πρέπει να βοηθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εργάτες και να λάβουμε υπόψη την παροχή βοήθεια προς 250 υπαλλήλους της εταιρείας αυτής. Μάλιστα, υπέρ λοιπόν. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. Η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κάποιος θέλει να ελέγξουμε την 20. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ για την 20. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 ε, κατά 11 υπέρ. Μία αποχή. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της εκθέσης. Α, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, τα citations στις ατολογικές αναφορές. Ξεχάσαμε. Η τροπολογία υπερθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η πέντε υπέρ κατά υπέρ λέω κατά άποχες απορρίπτεται και τώρα Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Next is... Um, E Επόμενα θέματα, κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων και η κυρία Γκαρτία Σαμπάλ είναι η συγγήτρια. Δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο ωστόσο και έτσι περνάμε στι ψηφοφορίε. Η τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Πάλι παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Θα σας ελέγξουμε αφού το επιθυμείτε. Έναρξη. Για την τροπολογία υπαριθμών 18. Πέρας. Απορρίφθηκε. 14 υπέρ, 14 κατά. Α, συγγνώμη, 15 υπέρ. Ήταν υπέρ ο κύριος Γκάιερ που δεν έχει την κάρτα του μαζί, άρα εγκρίνεται. Η 19 σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έγκρινεται. Η 20, 20 καταπίπτει, η 21 επίσης καταπίπτει. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες έγκρινεται. Τροπολογία 30. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε νοριακό. Την 37. Ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε 14 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. 15 υπέρ μάλλον με τον κύριο Γκάιερ. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την τρία. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. Η τέσσερα. Υπέρ. Καταπίπτει. Καταπίπτει τέσσερα, άρα η πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η έξι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η επτά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η εννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δώδεκα Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της χρηματοδότησης αποστροποποιήθηκε έναρξη, παρακαλώ. 21 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, 22 μάλλον υπέρ, 5 κατά, 2 εποχές. Next is implementation report on implementation report on Creative Europe. Rapporteur is Madam Moody. Η συγγήτρια δεν θέλει το λόγο. Θα ξεκινήσω με την δύο, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή.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 Πρέπει να ξαναξεκινήσουμε παρακαλώ την ψηφοφορία. Για ξαναψηφίστε παρακαλώ για την ε, τροπολογία 2. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε παρακαλώ και αυτήν. Ψηφίζουμε. Πέρας. 13 υπέρ, 12 κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται. γκρίνεται. Η 3 ήταν αυτή. Η πέντε τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας παρακαλώ να σηκώνετε καλύτερα τα χέρια σας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η επτά, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η έξι, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η οκτώ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Η 11. Διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Καταπίπτει, καταπίπτει. Η 10 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Η Ευρώπη για τους πολίτες τώρα. Ο κύριος Χριστοφόρου, ο εισηγητής. Που δεν είναι παρόν. Η τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος τότε για την 5 Ψηφίζεται. It has been rejected 15 to 12. Απερίφθη. 15 κατά 12 υπέρ. 7 υπέρ. συγγνώμη, οι δύο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Θέλετε να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάμε, ψηφίζετε για την 2. Δεκτή 15 υπέρ 12 κατά μία αποχή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή Επτά υπέρ κατά αποχές δεκτή Οκτώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη Εννέα υπέρ κατά αποχές απερίφθη Δέκα υπέρ κατά αποχές απερίφθη δώδεκα υπέρ κατά αποχές απερίφθη ένδεκα υπέρ κατά αποχές απερίφθη Δεκατρία υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Δεκατέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δεκαπέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 16 υπέρ. Όχι, δεν έχει καταπέσει. 16 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 16. Ψηφίζεται. Τέλος, δεκτή. 15 υπέρ 12 κατά. Ή 17 υπέρ κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. 19 και 20 ταυτόσημες υπέρ κατά. Αποχές απερίφθησαν. 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. «22» ξαναλέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές δεκτή. «23» υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24, 25, 26 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκ, απερίφθησαν προφορική 1 του εισηγητή ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ή μάλλον διορθώνει ο πρόεδρος δεκτή 27 Α, τότε θα ελέγξουμε την 27 τώρα. Ψηφίζεται. So it was rejected 15 to 11. Thank you for that. Ευχαριστώ. Περνάμε στην 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 29 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 30 και 31 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθησαν. 33 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 32 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36 υπέρ έχει καταπέσει 36, 37 τότε, 37 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. Ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία για το τροπολογημένο ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας δεκτή. 21 υπέρ 5 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, σε όλους τους εισηγητές. Το 14 τώρα στην ημερήσια διάταξη για τις μεταφορές. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Ο κύριος Φερνάνδης έχει το λόγο, παρακαλώ. Για τις μεταφορές, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια τη μεταφοράς ε, υπαριθμών 31, 856.800 ευρώ για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που μόλις ψηφίσαμε, που μόλις εγκρίθηκε. Μιλάμε για ένα ποσό δεσμεύσεων που ανταποκρίνεται στην οικονομική συνεισφορά. Ζητώ λοιπόν την έγκριση αυτής της μεταφοράς. to want to do Θέλετε να το δούμε ξεχωριστά αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, να ψηφίσουμε λοιπόν επ' αυτού ηλεκτρονικά. One more vote. Okay. The vote is closed. It's approved. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται και το 36 ναι. Το 36 είναι έτοιμα μεταφοράς 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για πληρωμές είναι για το όργανο που συνσφέρει σταθερότητα και στην ειρήνη και πάει προς την, στο όργανο σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια. Ζητώ λοιπόν την έγκριση και αυτής της μεταφοράς Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται λοιπόν 17-2 μία αποχή. 37-38-39 ναι. Βεβαίως οι μεταφορές 37-38 και 39 μαζί αφορά την, ένα ποσό συνολικά 85 εκατομμυρίων ευρώ για δεσμεύσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ιορδανία για τους Σύριους πρόσφυγες 20 εκατομμύρια προς το Τσάντ μετά την ξηρασία και τις ε, μετατοπίσεις 42 εκατομμύρια και ε, επίσης 25 ε, εκατομμύρια για τους εκτοπισμένους μετά την επίθεση κατά του Ισλαμικού κράτους στη Μοσούλη. Θα ήθελα να πω καλή τύχη ο Βιτζάι Πάτσα Watts, δεν ξέρω αν λέω καλά το όνομά του, θα μας αφήσει ο γραμματέας για το θέμα αυτό, διότι και αυτός εξαιρετείται την αξία της συνταξή του, θα μας αφήσει στο τέλος του μήνα να τον ευχαριστήσουμε λοιπόν για τη δουλειά του. Μάλιστα, άρχιτη ψηφοφορία. Και για τα τρία λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Λοιπόν, άλλα τμήματα. Ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρώτη μεταφορά αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο C8 2016 συλλέξαμε όλα τα ποσά τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί 53,5 εκατομμύρια ε, όπως και τα άλλα έτη δηλαδή το 2015 είχαμε 71 εκατομμύρια 71,5 το 2015 53 εκατομμύρια το 2016 όλα αυτά θα αφιερωθούν ε, στην, για την πληρωμή του ε, κτηρίου Κόνραντα Ντενάουερ. Δεν έχω κάποια αντίρρηση και προτείνω έγκριση. Εντάξει, ηλεκτρονικά ας το κάνουμε αυτό. Ο κύριος Μόνκερ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ βεβαίως αυτής της μεταφοράς δεν έχουμε και άλλη εναλλακτική, αλλά κατά, την, ε, κατά το σχεδιασμό του προπολογισμού είχαμε πει ότι γνωρίζαμε ότι αυτό θα ήταν γύρω στα 70 εκατομμύρια. Τώρα όμως ε, έχουμε 53,5 εκατομμύρια και έχουμε εγκρίνει και άλλα ποσά 150 εκατομμυρίων υπάρχουν μεταφορές ε, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Προεδρείο κατευθείαν. Βεβαίω έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, αλλά έτσι ε, δεν έχουμε διαφάνεια. Αυτή η προσέγγιση δημοσιονομική δεν είναι σε κανένα περίπτωση διαφανής. Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε στις, στα project αυτά έγκαιρα στις μελλοντικές μας, στο μελλοντικό μας σχεδιασμό να μπορούμε να εξοικονομούμε και χρήματα χωρίς να πληρώνουμε τόκους. Εάν το κάνουμε με μεγαλύτερη διαφάνεια, σίγουρα θα εξοικονομήσουμε περισσότερα. Διότι δεν είμαστε και μοντέλο σε ό,τι αφορά και παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά το υποσυνόμικο σχεδιασμό. Άλλα σχόλια πριν ψηφίσουμε. Ωραία, ας ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 18-2 μία αποχή. Λοιπόν, το επόμενο, η επόμενη μεταφορά, κυρία Ντεπρέ, ναι, Πρόεδρε, για το δικαστήριο ENF 8 2016 2,5 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις που, από τις αποζημιώσεις που μεταφέρονται στις αγορές και αυτό διότι ένας δικαστής ε, δεν πρόκειται να λάβει τα καθηκοντά του πριν το τέλος του έτους και έτσι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ε, την επέκταση ε, των κτηρίων του δικαστηρίου. Δεν ξέρω καν να πρέπει να ψηφίσουμε από αυτό. Δεν ξέρω, έχει κανείς αντίρρηση. είμαστε στα όρια των μεταφορών ε, πιστώσεων. Ε, δεν υπάρχει αντίρρηση, οπότε εγκρίνεται το επόμενο τώρα, το ελληνικό συνέδριο V 13 κάθετος 16 320.000 ευρώ μεταφορά για τη χρηματοδότηση ενός νέου project που λέγεται το μοντέλο εγγράφου της CEA για 136.000 ευρώ ε, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα έλεγα να μην φέρουμε αντιρρήσεις. Ε, ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε από αυτού. Εγώ θα ρωτήσω παρόλα αυτά αν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Ωραία, συνεχίζω. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προτείνει μια συνολική μεταφορά 1.300.000 ευρώ που προέρχονται από τις αμοιβέ ε, τους μισθούς για να, μεταφερθούν στη γραμμή που έχει να κάνει με τη βελτίωση της κρυπτογράφησης των επικοινωνιών για την ε, βελτίωση δηλαδή της ενίσχυσης της συνεργασίας ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι πολύ σημαντική για την προστασία εξωτερικής δράσης. Εγώ δεν έχω κάποια αντίρρηση. Φαντάζομαι ότι αν δεν έχουν και οι υπόλοιποι αντιρρήσει, ε, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Εντάξει, εγκρίνεται το επόμενο, τελευταίο. Η Επιτροπή Περιφερειών εδώ, τροποποίηση του σχεδίου ε, εγκατάστασης, ε, τέσσερις μόνιμες θέσεις αντέ 6 μετατρέπονται σε προσωρινές θέσεις αντέ 6 σεβόμαστε το άρθρο 50 των εφαρμοστέου κανόνα σε ό,τι αφορά το προσωπικό, οπότε προτείνω να το εγκρίνουμε. Αυτό δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτό. Το τελευταίο θέμα που θα εξετάζαμε αφορούσε την κτηριακή πολιτική, αλλά δεν υπάρχει έτοιμα για να συζητηθεί αυτό, οπότε ολοκληρώσαμε με τις ψηφοφορίες. Υπάρχει ο κοινός δημοσιονομικός έλεγχος τώρα. Ε, στις 12 είναι να γίνει η συζήτηση αυτή από κοινού με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, οπότε έχουμε μια διακοπή έως τις 12. Ευχαριστώ. je, non, non, non,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

Okay.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

No, no,

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

No me preocupa que,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 Καλώς ορίσατε στην κοινή συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμού και της Επιτροπής ε, Ελέγχου Προϋπολογισμών και αντιμετωπίζουμε σήμερα και πραγματευόμαστε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζητήμα, τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την αναθεώρηση του κανονισμού και θα δώσω πάρα αυτά το λόγο στην Συμπρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου την κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κοινή αυτή συνεδρίαση, την οποία στο μέλλον θα διεργανώνουμε και πιο συχνά. Καθότι και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε για το άρθρο 55 του κανονισμού βάσει του 55, θα καταρτήσουμε μία έκθεση. Εγώ θα είμαι από την Επιτροπή μας και ο συνεισηγητής ε, από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών θα αναλάβει τα δικά του καθήκοντα. Στην παρούσα λοιπόν φάση θα θέλαμε να πούμε ότι στη διάσκεψη του Προέδρου στις 22 Νοεμβρίου αποδέχτηκε την πρόταση των δύο επιτροπών σε ό,τι αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναρμόδιων επιτροπών και αποδέχτηκε λοιπόν ε, ε τη διαδικασία που προτάθηκε και θα μνημονευτεί και θα καταγραφεί και σε ένα μνημόνιο συνεννόησης. Και η ΙΤΡΕ ζήτησε συναρμοδιότητα σε θέματα όμνιμπους μόνο. Η τελική ε, εκδοχή και το τελικό σχέδιο της, ε, του μνημονίου συμφωνίας αυτής θα ε, δημοσιευτεί στα χέρια της γραμματείας. Και έχουμε και το Μνημπούς το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα. το κανονισμό που βασίζεται στο, άρθρο 55 στην αρμοδιότητα των δύο επιτροπών και το δεύτερο τμήμα αλλαγές 15 κανονισμών ανάλογα με τις μεμονωμένε κατηγορίες. Εμείς λοιπόν έχουμε ρέγγι, άγκρι, ίντρε και τραν στο πρώτο τμήμα, συνδεδεμένε. Ε, βάσει του άρθρου 54 και θα επεξεργαστούν τα τμήματα του μνημάς που υπάρχουν στι θερμοδιατητές του. Οι, λοιπόν, οι επιτροπές λοιπόν αυτές σε σχέση και με το άρθρο 54 και τα όσα προβλέπονται έχουν κάποια επιπρόσθετα δικαιώματα, πέρα δηλαδή από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 54. Είναι ε, αποκλειστική η αρμοδιότητά τους για τα τμήματα και του τομεί που είναι αρμόδια, δηλαδή θα περιμένουμε και θα ε, λάβουμε υπόψη και θα αποτεχτούμε χωρίς ψηφοφορία τις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών αυτών. Στο δεύτερο τμήμα τώρα των αρμοδιοτήτων, θα γίνουν ε, αυτόνομα και παράλληλα η ε, τριμερή διάλογοι παράλληλα προς την Στρελόκουσα ε, με και το πρώτο τμήμα. Θα συναντιόμαστε τακτικά, θα υπάρξει και ένα coherence forum, ένα forum συμβατότητας και ομοιογένειας και θα συμμετέχουν όλοι οι πρόεδροι των αρμόδιων επιτροπών γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ομοιογένειας. Ο Πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και η, πρόεδρο η πρόεδρος ε, του, της Προπολογισμού και η πρόεδροι των των επιτροπών ε, θα συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή. Θα προσπαθήσουμε να συντονιστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και επιπλέον βάσει του άρθρου 53 θα καταφυστούν και εκνομοδοτήσεις οι οποίες και θα ψηφιστούν στις ε, αρμόδιες επιτροπές και η Επιτροπή ε, Προπολογισμού και Ελέγχου των Προπολογισμών μπορούν να λάβουν υπόψη τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Ως Έχουμε μόνο ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας με την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Το Coherence Forum θα λάβει για πρώτη φορά χώρα την επόμενη Δευτέρα. Όποιος θέλει να έρθει. Να Και έχουμε και κάποια προσωρινά στοιχεία, έτσι, για προσανατολισμό. Έχουμε τέλη Φεβρουαρίου ένα εργαστήριο, καλέσαμε και την Επιτροπή Ευλέγχου Προπολογισμού, 2 Μαρτίου, ε, τέλη Μαρτίου περιμένουμε να μεταφραστεί το κείμενο και να συζητηθεί το θέμα τέλη Μαρτίου στις Επιτροπές και μετά θα έχουμε άλλη μια κοινή ε, συνεδρίαση. Αρχές Μαΐου η κοινή ψηφοφορία θα λάβει χώρα. Ελπίζουμε οι τριμερείς διάλογοι μέχρι το θερινό διάλειμμα να μπορέσουν να έχουν ολοκληρωθεί. Αρχές Σεπτεμβρίου το συμβαστικό κείμενο, αν όλα έχουν πάει καλά. Θα ψηφιστούν στις δύο επιτροπές ελέγχου προπλογισμού και προπλογισμού και μετά θα αρχίσουν να ισχύουν από 1η Πρώτου 18 οι νέοι, ο νέος κονισμός. Θα αρχίσει να ισχύει τον Ιανουάριο του 2018 η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την επόμενη αναθεώρηση. Συνεχίζονται λοιπόν ε, οι μεταρρυθμίσει και οι αναθεωρήσει. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξο το σχεδιάγραμμα αυτό. Φυσικά το ξέρουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα για να πετύχουμε το οτιδήποτε στην παρούσα φάση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από όλε τι ε, εμπλεκόμενε επιτροπέ να κάνω γρήγορα η όλη διαδικασία ασφαλώς ε, θα αποτελέσει δοκιμασία για τις διάφορες ε, επιτροπές ε. και υπάρχει πειρασμός φυσικά να καταθέσει κάθε επιτροπή 2.000 τροπολογίες. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ο πειρασμός αυτός, αλλά ας προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Αν θέλουμε να έχουμε κάποια επιρροή στην παρούσα περίοδο, την προγραμματική περίοδο, ε, ο χρόνος θα παίξει σημασία. Πώς θα το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα αυτά. Γιατί θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να κάνει πίσω σε προτάσει απλοποίηση. και να πάρει και ο συνάδελφος, ο Ρίτσαρτ, το λόγο για να μας μιλήσει ως συνεισηγητής. Uh, <coughs> Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι συνεισηγητής. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή του Ελέγχου που μου ανέθεσαν αυτό το έργο. Κάποια σχόλια για να υποστηρίξω αυτά που είπε μόλις η Πρόεδρος. Έγινε αναφορά στο γεγονός ότι πολλές επιτροπές θα έρθουν να συνεισφέρουν στο θέμα αυτό. Είναι περίπλοκο λοιπόν το εγχείρημα και ανέφερε πώς σκοπεύουμε, πώς προτείνουμε να συνεργαστούμε με τρόπο συνεκτικό. Αλλά βέβαια ο εχθρός θα είναι πάντα ο χρόνος. Έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης έως το καλοκαίρι, είναι φιλόδοξο αυτό, είναι εφικτό, αλλά θα εξαρτηθεί από την καλή θέληση και τη συνεργασία όλων όσων ε, θα συμμετάσχουν. Κάνω λοιπόν έκκληση και σε εκπροσώπους άλλων επιτροπών να αντιληφθούν ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και θα χρειαστούμε βοήθεια από παντού. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αν υπάρχει μια θεματική η οποία ε, επανέρχεται συχνά στη συνεισφορά μου ε, είναι η απλοποίηση. Ξέρω ότι πρόκειται για μια εμβληματική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή και εμείς το ενθαρρύνουμε αυτό και το καλωσορίζουμε. Ο κίνδυνος είναι όμως να μπλέξουμε, να μπλέξουμε τις λεπτομέρειες και να χάσουμε την ευρύτερη εικόνα, τον ευρύτερο στόχο θα ήθελα λοιπόν όσοι όσοι συνεισφέρουν να το λάβουν υπόψη αυτό. Βεβαίως αναμένουμε συνεισφορές των ε, συναδέλφων για το πώς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και αναμένω με ανεπιμονησία τη συνεργασία με την Ίγκη για να φτάσουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δύσκολο να πετύχουμε θέματα απλοποίησης είναι τόσο περίπλοκο ζήτημα και στην ανάγνωση του πρώτων αρθρών δεν μπορούμε να πούμε ότι από πλευρά διατύπωση τα πράγματα είναι πιο απλά και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διάθεση να επεξεργαστεί εκ νέου κάποιες διατυπώσεις. Έγινε και μια πρώτη συνάντηση με την Επιτροπή. Κάναμε κάποιες παρατηρήσεις, τις πετάξαμε από πάνω μας. Προέκυψαν και κάποια non-paper. Νομίζω ότι ακόμα και καταφέρουμε να γλιτώσουμε από τον αρμόδιο υπάλληλο το να διαβάσει το κείμενο πολλαπλέ φορέ μέχρι να το καταλάβει, θα ήταν μια απλοποίηση. Αυτά, Πρόεδρε, από πλευρά μου, αυτή ήταν η δική μου παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ε, και ταυτόχρονα συνεισηγήτρια. Λοιπόν, τώρα θα έχω μια ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος Μόγκ και Μάνκα έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω για τη διαδικασία αλλά και για κάποια επιμέρους ε, ουσιαστικά ζητήματα. Εάν θέλουμε να εξοικονομήσουμε, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων, είναι κάτι το οποίο συζητάμε και εδώ και χρόνια, έτσι. Θα πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα θεσμικά όργανα. Και αν δεν δοθούν κίνητρα, ε, δεν θα υπάρξει εξοικονόμηση. Αν υπάρχει κάποια δυνατότητα πλεονασματική σε ένα θεσμικό όργανο, ε, θα πρέπει να διατίθεται αλλού και θα πρέπει βεβαίως να δίνονται και κάποια κίνητρα για να συμβεί αυτό. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα τώρα, η Επιτροπή Ρέγγιο και η Επιτροπή Άγκρη σίγουρα θα χρειαστούν πολύ χρόνο. Δεν νομίζω ότι θα ολοκληρώσουν τις θέσεις τους ε, έως τα τέλη Ιανουαρίου. Γιατί δεν τους δίνουμε άλλο ένα μήνα για να προλάβουν. Κάτι άλλο τώρα. Η απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων σίγουρα θα συνεισφέρει στη μείωση του κόστους. θα μας επιτρέψει να κινηθούμε πιο γρήγορα και με λιγότερα λάθη. Πρέπει όμως ε, να μελετήσουμε ποιοι είναι οι λόγοι για την αργή εφαρμογή. Ε, διότι αυτό δημιουργεί τεράστιες απώλειες και σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και σε επίπεδο απασχόλησης. Πρέπει αυτό ε, να το μελετήσουμε. η απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί και με τη μείωση των επιπρόσθετων επαληθεύσεων. Νομίζω δεν χρειάζονται τόσες επαληθεύσεις, τόσοι μηχανισμοί ελέγχου. Και αυτό θα οδηγήσει, θα οδηγήσει εξοικονόμηση και αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξετάσουμε, να γίνουν μελέτες, ε, να δούμε κατά πόσο αυτές οι επαληθεύσεις, οι, επαληθεύσεις, οι έλεγχοι, οι ex post είναι αποτελεσματικοί ή όχι, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία για αυτά. Το ποσοστό ε, ευρημάτων μπορεί να είναι τόσο μικρό που το κόστος της όλης διαδικασίας να είναι μεγαλύτερο από τα όποια ωφέλη προκύπτουν. Τώρα ο συνδυασμό ε, χρηματοδότηση από τα ταμεία, τα διαφορετικά και τα ταμεία, τα επενδυτικά και από το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο. Ε, ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων είναι ένα συμπληρωματικό ταμείο. Ε, ο λόγος ύπαρξής του είναι να διαθέτει κονδύλια όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα χρηματοδότησης. Αυτό επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να παράσχει κάποιες εγγύησεις. Δεν ξέρω όμως αν η προσέγγιση της Κομισιόν αυτή είναι η κατάλληλη, δηλαδή να βρεθούν χρήματα και από τα δύο ταμεία. Δεν μπορώ να το ε, συλλάβω ακριβώς πώς θα συμβεί αυτό. Στο επταετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, κατά την προσπάθεια αναθεώρησής του, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε πλεόνασμα προκύψει κατόπιν κάποια κύρωση που έχουμε επιβάλει, παραδείγματο χάρη, πρέπει αυτό το πλεόνασμα να μπορέσουμε να το ε, διατηρήσουμε χωρί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε τι συνεισφορέ των κρατών μελών. Είναι και αυτό. Είναι πολλά τα εκκρεμή ζητήματα. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε πιο λεπτομερώ, να συζητήσουμε και τη διαδικασία. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να ε, διευρυθεί κάπως το χρονοδιάγραμμα για να έχουν τον χρόνο οι άλλες επιτροπές ε, για να συνεισφέρουν επικοδομητικά, όπως η Ρέτζιου και η Άγκρη. Ο κ. Γκάιερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πολλή εμπειρία για το θέμα αυτό. Την τελευταία φορά όμως όταν το κοιτάξαμε, ήμουν σκιώδης. Και ο κύριος Μιλτερ το ανέλαβε από τους φιλελεύθερους και Πέρασαμε κάποια χαρούμενα απογεύματα με τις άλλα ε, θεσμικά όργανα για να αντιπραγματευτούμε τα όσα μας απασχολούσαν. Δεν το έχω εξετάσει σε βάθος το θέμα ακόμα, αλλά μια πολιτική εκτίμηση θα ήθελα να ζητήσω σε αυτή τη φάση. Σε τι βαθμό λοιπόν τα παλιά προβλήματα, οι παλιές επιθυμίες αν θέλετε του Κοινοβουλίου και τα εντοπισμένα προβλήματα ανακύπτουν και πάλι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν λεφθεί υπόψη αυτά που έχουμε πει και έχεις οποιαδήποτε ένδειξη για το τι προθυμία ε, δείχνει το Συμβούλιο στην παρούσα φάση. Θυμάμαι και τη συζήτηση που έγινε για τα δημοσιονομικά μέσα, τα οποία ήταν πολύ περιορισμένα. Τώρα έχουμε κάποια χρόνια εμπειρία πλέον, επαρκή εμπειρία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο υπέροχα όσο μας έλεγαν το 2013 και 2014 και σε ό,τι αφορά τον πώς λειτουργούν τα πράγματα και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, το χρηματοοικονομικό. Ερωτούμε λοιπόν ε, κατά πόσον είναι σωστή η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύεις ότι σωστά ανταποκρίνεται σε όσα ζητήσαμε και χρειαζόμαστε. Και το Συμβούλιο έχει πρόθεση και διάθεση να διαβουλευτεί. Ύστερα έχουμε και τους ε, δορυφόρους της, ε, του προπολογισμού που δεσμεύουν αφενός τα ευρωπαϊκά μέσα από την άλλη, εκνευλευτικό έλεγχο για την ε, χρήση των κονδυλίων αυτών μειώνεται. Τρίτη ερώτηση. Budget for results. Το έβαλε αυτό και το έθεσε θέμα η Κρυσταλίνα Γεωργίευα, το θέμα της ενέργειας για τη βελτίωση της απόδοσης. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο αποτυπώνεται στο σχέδιο όμως του προπολογισμού. Και κάτι άλλο που απασχολεί ιδιαίτερα πάντα το Κοινοβούλιο, το θέμα της λογοδοσίας των κρατών μελών. Έχουμε ταπανίσει πάρα πολύ ενέργεια, αλλά με περιορισμένα αποτελέσματα. Θα το βάλουμε λοιπόν το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, σε κάποια φάση. Ε, εγώ θα ήμουν υπέρα, αλλά δεν ξέρω και αν αξίζει και τον κόπο. Διάφορε ερωτήσει, λοιπόν απευθύνθηκαν προ την εισηγήτρια. Δεν ξέρω αν θα θέλεις να απαντήσεις. Α, ας ακούσουμε τον κύριο Τάραντ όμω πρώτα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα των κανόνων που θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι και κυρίως απλούστεροι. Στα πλαίσια αυτής της περίπλοκης διαδικασίας των πολλών επιτροπών που εμπλέκονται και των πολλών οργάνων, να μην ξεχνάμε επίσης και την ε, Give all participants in the process equal rights. They serve us. Θα πρέπει να υπάρξει ισοτιμία για όλους, θα πρέπει να είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο απέναντι στις ρυθμίσεις αυτές. Γι' αυτό θα στηρίξω τους δύο εισηγητές στην προσπάθειά τους να απλουστεύσουν και να διασφαλίσουν ένα ισότιμο πεδίο ε, εφαρμογής του τελικού προϊόντος. Προσπαθώ να συμμετέχω στη διαδικασία αυτή όσο περισσότερο ε, οι άνθρωποι της Επιτροπής Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού πολλές φορές ε, είναι το ίδιο πρόσωπο. Και γι' αυτό η λεπτομέρεια έχει σημασία ε, όταν βάλεις το, στη σωστή θέση το κόμμα τότε δεν θα πρέπει να το κάνουμε σαν τον Τσέγκης Χάν, ο οποίος έγραψε pardon not to be executed, αλλά ξέχασε να βάλει το κόμμα και εκτελέστηκαν οι στρατηγοί του. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο θέλω να υπογραμμίσω, το οποίο θέλω να υπογραμμίσω. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι εφικτό. Είναι οι διαδικασίες ελέγχων αν θέλετε που θα πρέπει να ακολουθούν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε επίπεδο διοικητικό. Είναι ένα μήνυμα που προέρχεται επίσης και από τους γεωργούς σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει εμείς στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης ε, να κάνουμε κάτι το πολύ συγκεκριμένο, γιατί αλλιώς δεν θα πω ότι αποτύχαμε, αλλά σίγουρα δεν θα έχουμε κάνει τη δουλειά μας. Αυτό θα ήθελα να προσθέσω. Ίσως η κυρία Γκρέσλε θέλει τώρα να δώσει κάποιες απαντήσεις και μετά από αυτήν ο κύριος Άσουερθ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Κοιτάξτε, να μετριάσουμε και λίγο τις προσδοκίες μας. Με την ε, μεταρρύθμιση αυτή και με την Omnibus θα επιλύσουμε κάποιες λίγες, ε, κάποια λίγα προβλήματα. Δεν πρόκειται να ε, κάνουμε στην ολική αναθεώρηση του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια μόνο ζητήματα θα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε κάποιες ε, μεγάλες αντιφάσεις του κανονισμού μας ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν τέτοιες μεγάλες αντιφάσεις. Αυτά προσπαθούμε κάπως να τις απαλύνουμε, κάπως να τις επιλύσουμε. Το κατά πόσο θα τα καταφέρουμε τώρα δεδομένου και του μορφότυπου που επιλέξαμε αναγκαστικά στην παρούσα φάση, δηλαδή με μεγάλη ε, απολυστική αρμοδιότητα των επιτροπών, δεν ξέρω, γιατί δεν έχουμε και δυνατότητα παρέμβαση σε τελική ανάλυση. Μην τα ανατρέψουμε και όλα, γιατί πολλά έχουν αποδείξει την αξία τους. Στην παρούσα φάση, στο Omnibus, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο show, road show από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξυπνά μεγάλε προσδοκίε, οι οποίε ω τώρα δεν μπορώ να πω ότι απαντώνται στο κείμενο. Και να πάω προ τον κύριο Μάνκα ότι οι επιτροπέ ασφαλώ θα έχουν το ίδιο χρονοδιάγραμμα με εμά. Και αυτοί μέχρι τέλη Μαρτίου πρέπει να έχουν τελειώσει. Μέχρι το Μάρτιο έχουν το χρόνο του. Δεν είναι και τόσα πολλά όπω ε, εμεί. Ε, γιατί εμεί τελικά είμαστε οι χαζοί και οι χαμένοι. Έχουμε τεράστιο όγκο να επεξεργαστούμε και να διαβάσουμε. Και εμεί έχουμε το πιο, το πιο λίγο χρόνο. Ε, οι επιτροπέ σε σχέση με το τομέα αρμοδιότητάς τους, καλό χρόνο έχουν. Θα προσπαθήσω να τα βγάλω πέρα, τι να σα πω, μαζί με τον Ρίτσαρτ. Αλλά δεν θα είναι εύκολο, σα το λέω. Ο Γιάννη τώρα, ο κύριο Γκάιερ. Έθεσε εκ των κάποια ερωτήματα και το εκτιμώ αυτό. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε λοιπόν είναι το εξή. Ε, για να απαντήσω και στον κύριο Μανκά, έχουμε λιγότερου ελέγχου. Ναι, λιγότερου ελέγχου, αλλά εμεί θέλουμε πιο αποτελεσματικού ελέγχου. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Το στην συνέδριο συνέχεια τι λέει, ότι δεν είναι αποτελεσματική η ελέγχή μα. Και τι νόημα έχει να κάνουμε πολλαπλού μη αποτελεσματικού ελέγχου. Άρα, θα πρέπει να δούμε το accountability chain, αυτή την αλυσίδα λογοδοσία, να αλλάξει με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να υπάρχει η αποτελεσματικότητα που θέλουμε. Και τελικά τι γνώσει που έχει ο καθένα να μπορεί να τι εφαρμόσει σε συγκεκριμένα μέτρα. Ε, αυτό ελπίζω να πετύχουμε με όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε πλέον. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Και yes, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τα Provisional 12. Εμείς είχαμε πει ότι είχαμε τρία ζητήματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντιταχθεί και τώρα έχει προσθέσει άλλα 12 σημεία. Το επέκτηνε λοιπόν αυτό. Πολύ. Γιατί δεν ξέρω. Να το συζητήσουμε. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να συμπεριληφθούν τόσα πολλά σημεία. Για τα χρηματοοικονομικά μέσα βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων έχει γίνει δουλειά για την πιο καλή και πιο ομοιογενή διαμόρφωση των ε, ε, εκθέσεων αυτών. Αυτό όμω ξεκίνησε από μια αρκετά άσχημη κατάσταση. Ήταν πολύ ε, μεγάλα τα προβλήματα. Τώρα λοιπόν έχουμε κάποια πιο ομοιόμορφη διαμόρφωση, να δούμε όμω ποιε θα είναι συγκεκριμένε προτάσει και ποια συνέπειες θα έχουν οι προτάσεις αυτές. Εγώ τι εντύπωση έχω, ότι κάποια μέτρα του κανονισμού έχουν ληφθεί για να μπορούν να τα παράνται πιο εύκολα τα χρήματα. Αλλά βασικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τους διεθνείς οργανισμούς. Εδώ λοιπόν θα μειωθούν οι υποχρεώσεις ελέγχου για τους ελέγχους που ορίζονται από τα διεθνή όργανα κτλ. Αυτό μπορώ να το αποδεχτώ. Αυτό που δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι όταν έχουμε λόγο να εξετάσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή όταν υπάρχουν σκάνδαλα, να υπάρχει αυτή η υποχρέωση λογοδοσίας των κρατών βελτίωση των υπηρεσιών διεξαγωγή των ελέγχων και στο ΕΦΣΥ τα ξεχωριστά θέματα. Το θέμα των δορυφόρων. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί εκ νέου το θέμα του ποιε είναι οι επιπρόσθετες, ε, τα επιπρόσθετα δημοσιονομικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να έχει σίγουρα απαντήσει σε ένα τμήμα των αξιώσεών μας, όχι σε όλες όμως και ενδεχομένω ε, να υπάρχει και ζήτημα σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και θα χρειαστεί σίγουρα και το αναλόγο χρονικό διάστημα. Mr. <clears throat> Ναι, ναι, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια τα οποία βρίσκω εξαιρετικά χρήσιμα. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα ε, στο σχόλιο που μόλις αναφέρθηκε ε, όντως μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στο να διαχειριστούμε τις προσδοκίες. Ε, δεν πρόκειται εδώ να αλλάξουμε τα πάντα και να επανεφεύρουμε όλο το σύστημα, προφανώς. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι αφενός να συνεισφέρουμε στο να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στους κανόνες και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της διαδικασίας προπολογισμού εδώ, αλλά και δημιουργώντας ένα, μια μέθοδο φιλική προς το καταναλωτή, αν θέλετε, στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι φορά το θέμα της απλοποίησης, και εδώ συμφωνώ απόλυτα με την Πρόεδρο, το ίδιο ακούω και εγώ από τους γεωργούς. Ε, είμαι και ο ίδιος γεωργός, το ακούω και στην οικογένειά μου κάθε Σαββατοκύριακο. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ευκολότερη πρόσβαση, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχει μια αίσθηση αναλογικότητας. Όλα αυτά με βρίσκουν σύμφωνο. Αλλά προσοχή, διότι πρέπει να βρεθεί ένα σωστό σημείο ισορροπίας. Ανάμεσα σε αυτό που είναι εύκολα προσβάσιμο και αυτό που είναι υποχρεωτικό. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή, να έχουμε ε, χαμηλά επίπεδα συμμόρφωσης και τελικά να διαπιστώνουμε ότι έχουμε οπισθοδρομήσει. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένα σημείο ισορροπία το οποίο είναι δύσκολο. Συμφωνώ πάντως σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε η πρόεδρος επ' αυτού. Η Γκάρ είπε κάτι ενδιαφέρον ε, σε ό,τι αφορά το budgeting. Το budgeting είναι καλό ή κακό ανάλογα με τους στόχου που έχει θέσει κανείς. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλαμε να πετύχουμε για να δούμε την απόδοση του προπολογισμού, το performance budgeting. Ε, και για το τελευταίο που είπατε, ο κύριος Μπάνκερς αναφέρθηκε στο θέμα το χρονικό, ότι πάντα ο χρόνος θα είναι ο εχθρός αυτής της έκθεσης. Ναι, εντάξει, λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά Άμα αρχίσουμε να δίνουμε χρόνο και παρατάσεις θα, θα τα πράγματα. Έχουμε φιλόδοξο στόχο. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε με το συνεισηγητή βέβαια για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ε, πραγματικά κάνω μια έκκληση ξανά για άλλη μια φορά σε όλες τις επιτροπές. Θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε να το κάνουμε έγκαιρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς, άλλα σχόλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να καλωσορίσω και να συγχαρώ την το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη γρήγορη αντίδραση. Θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο τώρα να κάνει το ίδιο, έτσι ώστε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε ένα εφικτό, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα καλά σχόλια που έγιναν. Θα ήθελα να αντιδράσω και εν συντομία σε κάποια από τα θέματα που τέθηκαν. Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ex post έλεγχοι αποτελεσματικοί. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα, όπου είναι εφικτό, ενιαίος έλεγχος, όπου είναι εφικτό βέβαια. Ιδάλλως βεβαίως πρέπει να διασφαλίσουμε τον, ε, το δικαίωμα στον έλεγχο. Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που ήθελα να αναφέρω στα πλαίσια και των συζητήσεων όπω εξελίσσονται στο Συμβούλιο. Είναι μια σημαντική πρόταση για την απλοποίηση, αλλά υπάρχουν δύο βασικοί στόχοι, έτσι. Ο άλλος στόχος είναι η ευελιξία. Η ευελιξία παραμένει σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκαμε εδώ σε κάποιες σημαντικές πτυχέ όπω η επαναχρησιμοποίηση των αιτήσεων δεσμεύσεων, ε, το θέμα του πλεονάσματο. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι εύκολε συζητήσει από ε, αυτών των θεμάτων, αλλά εμεί θα επιμείνουμε. Τώρα, όλοι αυτοί οι δορυφόροι, όπω του ονομάζουμε γύρω από τον προπολογισμό, προσπαθούμε αυτά να τα βάλουμε σε υπό ένα νέο τίτλο ε, ε, δημοσιονομικές οικονομική ενίσχυση θα δούμε αν θα γίνει αποδεκτό υπάρχει πάντως μια πρόταση για αναδιοργάνωση όλου αυτού του συστήματος και κάτι για, την, για τη διαχείριση, την κοινή διαχείριση και την λογοδοσία των κρατών μελών. Εμεί θεωρούσαμε ότι δεν ήταν, δεν ήταν σκόπιμο σε αυτή τη στιγμή να προτείνουμε σε βάθο μεταρρύθμιση τη μοιρασμένη διαχείριση. Είμαστε στα μέσα του προγράμματο. Καλύτερα να το αφήσουμε αυτό για το επόμενο πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο, όπου θα επανεξετάσουμε σε βάθο ε, αυτού του κανόνε. Προτείναμε βεβαίω κάποιε σημαντικέ βελτιώσει, όπω το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων και διευκρίνηση των σχετικών κανόνων. Τώρα και τα οικονομικά μέσα προσπαθούμε βεβαίως να βελτιώσουμε τους κανόνες, όχι να τους καταργήσουμε, να τους βελτιώσουμε χωρίς να χάνονται σημαντικές πληροφορίες. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οι διερμηνείς θα φύγουν, θα σταματήσουν σε ένα λεπτό. Οπότε ο παρακαλώ να είναι πάρα πολύ σύντομο, να είναι πολύ σύντομο, 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Θα ήταν καλό ε, πώς λέμε καλά Χριστούγεννα σε όλους, όλες τις γλώσσες, αφού είναι οι ακόμα εδώ. Καλά Χριστούγεννα. Πολύ ωραία. Η, τελευταία, η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα ενδεχομένω στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των συζητήσεων του Προέδρου και της εισηγήτριας ε, τη συνάντηση που έχουν στο Συμβούλιο σήμερα ε, οπότε υπάρχει και ένα ποτό της ομάδας ε, δημοσιονομικού ελέγχου με την Αντιπρόεδρο την κυρία Γεωργίευα με αφορμή την αποχώρησή της αυτό θα γίνει εδώ έξω από